11 η ώρα. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση του κυρίου Κάπουλας Σάντος. Κανονισμός ε, υπαριθμών ε, 73 και ποσοστό αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων προβλέπονται σε αυτόν όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2013. Ο εισηγητής, ε, κ. αν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε πίτροπε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, παρά τις προσπάθειες του Επιτρόπου Σιόλος για να έχει τον απαραίτητο προπολογισμό η Γεωργία, τελικά μέχρι το 2020 από το 2014 ο προπολογισμό της Γεωργίας θα είναι σοβαρά μειωμένος. Ήδη από το 2014 θα υποχρεωθούμε να εφαρμόσουμε το μηχανισμό δημοσιονομικής πειθαρχίας κατά πάσα πιθανότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ως βάση υπολογισμών την πρόταση προπολογισμού που είχε εγκριθεί από το Συμβούλιο στις 8 Φεβρουαρίου. Με αυτή τη χειρονομία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας εξέπληξε, μας ευνηδίασε και μας ανάγκασε να να αποδεχτούμε οριστικά τον προπολογισμό όπω τον είχε εγκρίνει το Συμβούλιο, αγνώντα τη διαδικασία συναπόφαση και όσα προβλέπει η συνθήκη τη Λισαβόνα. Η θέση αυτή δείχνει ελάχιστο σεβασμό προ τη Θεσμική Συμφωνία και το Ευρωκοινοβούλιο και βεβαίω εδώ εκφράζουμε τι έντονες επικρίσεις μα. Η εναλλακτική πρόταση που υποβάλαμε είναι αυτή που εγκρίθηκε με τη διαπραγματευτική εντολή κατά μεγάλη πλειοψηφία και με την έγκριση της Ολομέλειας περάσαμε στην συζήτηση για τον κανονισμό των άμεσων πληρωμών. Είναι η μόνη πρόταση που θεωρούμε αποδεκτή στην τωρινή συζήτηση στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Επίσης, πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει το μηχανισμό αυτό να μην τον εφαρμόσει στους γεωργούς που λαμβάνουν λιγότερο από 5.000 ευρώ το χρόνο. Ένα μεγάλος αριθμός των γεωργών, 80% περίπου του συνόλου, που λαμβάνουν μόνο 15% του συνολικού ποσού. Η θετική διακριτική μεταχείριση των μικρότερων και η στόχη της απλούστευση που είναι κάτι που διαρκώς ε, επικαλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάτι που δικαιολογεί τη στάση μας. Καλό λοιπόν την Ολομέλεια να εγκρίνει την έκθεση που σήμερα συζητούμε. Σας ευχαριστώ. Ο Επίτροπος Τσόλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ζηγητά. κύριε και κύριοι, η πρόταση που αφορά την εφαρμογή του δημοσιονομικής πειθαρχία την έκανε την πρόταση αυτή η Κομισιόν διότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας για τον προϋπολογισμό του 2014 δεν έχουμε αρκετή χρηματοδότηση για τα μέτρα διευθέτησης των αγορών. Και γιατί λοιπόν πήραμε υπόψη μας τα ποσά που προβλέπονται στις δημοσιονομικές προοπτικές του Συμβουλίου που ενέκρινε το Συμβούλιο δηλαδή και όχι αυτές που πρότειναμε εμείς αρχικά πολύ απλά για λόγους πραγματισμού. διότι δεν είχαν ακόμη εγκριθεί δημοσιονομικές προοπτικές και από το Κοινοβούλιο αλλά από τότε αποσαφηνίστηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ότι έπρεπε το Κοινοβούλιο να εγκρίνει και τώρα το διαπραγματεύεται αριθμούς που είναι πολύ μειωμένοι σε σχέση με τους δικούς μας. Για αυτούς τους λόγους ρεαλισμού και πραγματισμού λοιπόν και για να έχουν οι ένα μήνυμα πιο ρεαλιστικό θελήσαμε να αναφέρουμε τους αριθμούς αυτούς που προέρχονται από έναν από τους συνομοθέτες, δηλαδή το Συμβούλιο, με τον όρο βέβαια να εγκριθούν οι δημοσιονομικές προοπτικές και λέω με τον όρο διότι υποαίρεση, διότι η εφαρμογή αυτή της δημοσιονομικής πειθαρχία είναι υποχρεωμένη να την κάνει η Κομισιόν για να γνωρίζουν οι γεωργοί σε τι να βασιστούν το επόμενο έτος, αλλά υπάρχουν πάντα τρόποι να προσαρμοστούν οι προτάσεις αυτές με βάση κάποια απόφαση ή συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Όπως ξέρετε έχουμε τη συνήθεια το φθινόπωρο κάθε έτος να κάνουμε διορθωτικό προϋπολογισμό ή με διορθωτική επιστολή μάλλον αλλάζουμε τον προϋπολογισμό και αν μέχρι το φθινόπωρο συμφωνήσει το Συμβούλιο με το Κοινοβούλιο για τις δημοσιονομικές προοπτικές τότε θα μπορέσουμε να πάρουμε υπόψη μας τους τελικούς αριθμούς και να τους ε, εφαρμόσουμε. Αλλά για λόγους ρεαλισμού το λέω για τρίτη φορά προτιμήσαμε να πάρουμε αριθμούς πιο κοντινούς στην περίπτωση μιας συμφωνίας εφόσον επιτευχθεί. Αποφασίσαμε δηλαδή εξ άντε από την ε, τελική εφαρμογή να μειωθούν οι επιχορηγήσεις για όσους γεωργούς έχουν κάτω από 5.000 ευρώ. Αυτές οι άμεσες επιχορηγήσεις προβλέφθηκαν για να διευκολυνθούν οι υπολογισμοί και για τις πληρωμές που ξεπερνούν 5.000 ευρώ, μας φάνηκε δηλαδή λογικό, και για αυτούς που έχουν κάτω από 5.000 ευρώ το χρόνο να μην εφαρμοστεί αυτή η εξαίρεση των 5.000 ευρώ. Κάτι ανάλογο είχε προβλέψει η Κομισιόν και για την αναθεώρηση της κοινή αγροτικής πολιτικής για να διατηρηθεί αυτή η εξαίρεση και να προστατευθούν οι μικρομεσαίοι καλλιεργητέ. Αυτά σας τα λέω για να ξέρετε γιατί προτείναμε αυτή τη δημοσιονομική πειθαρχία και γιατί λάβαμε υπόψη μας μερικούς αριθμούς που θεωρούμε πιο κοντά σε μια πραγματικότητα ξαναλέω για να δοθεί ένα, για να καταλάβουν οι γεωργοί σε τι πρέπει να βασιστούν του χρόνου. Αλλά όλα αυτά με την αίρεση μιας έγκρισης των προοπτικών από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Αν φυσικά αυτή η απόφαση δεν υπάρξει καιρός τότε θα ισχύσουν οι κανονισμοί που μας υποχρεώνουν να εφαρμόσουμε άλλου είδους μηχανισμούς, άλλου είδους. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Και τώρα, για ένα λεπτό, ο κύριος Λαβία, από την Επιτροπή των Προπολογισμών. Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, ως εισηγητής για την έκθεση αυτή στην Επιτροπή των Προπολογισμών θα σταθώ στα δημοσιονομικά τμήματα τη έκθεση αυτή, όπω είπε ο επίτροπο, αλλά και ο εισηγητή. Θέλουμε να εγκρίνουμε, ή μάλλον έχουμε περάσει τις διαπραγματεύσει για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Τώρα όμω δεν ξέρουμε ακόμα τι πόρους θα διαθέτουμε και σε ποιε γραμμέ του προπολογισμού. Ξέρουμε ποιο θα είναι το μέγιστο όριο ε, που θα ισχύει για το 2014, αλλά και αυτό ακόμη δεν είναι απολύτω βέβαιο. Πριν οριστεί ένα το όριο λοιπόν, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορούσαμε να προσαρμόσουμε τι πληρωμέ που οφείλονται για το 2010. Είμαστε σκόπιμο άρα να προτείνουμε την αναθεώρηση του κανόνα για τη δημοσιονομική πειθαρχία. Και αυτό στην Επιτροπή Προπολογισμών και κατά τη διαδικασία έγκριση του προπολογισμού του 2014. Να σα θυμίσω, Επίτροπε, αυτό που είπατε και εσεί για τη διορθωτική επιστολή. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία για το ε, πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, κάτι που αυτή τη στιγμή δεν αποκλείεται, Πώς θα εφαρμοστεί η δημοσιονομική πειθαρχία εφόσον οι συνεισφορές θα υπολογιστούν στο ανώτατο όριο του 2013 με ποσοστό αύξηση 2% βάσει του πληθωρισμού. Πρόεδρος, ευχαριστούμε και τώρα για τρία λεπτά ο κύριος Γιάννη. Äh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Για το επόμενο έτος η Κομισιόν προβλέπει την περικοπή των άμεσων πληρωμών στους Ευρωπαίους αγρότες και θεωρώ ρεαλιστικό το να ασχοληθεί η Κομισιόν με τον προϋπολογισμό ο οποίος μειώνεται, αλλά ανεξαρτήτως αποτελέσματος πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός για το τι θα γίνει όταν ξεπερνάμε τον προϋπολογισμό. Έχουμε προβλέψει κάτι ανάλογο και στην κοινή οργάνωση αγοράς. Και Όσο κατανοητή και αν είναι η δημοσιονομική πειθαρχία, τόσο ε, κατανόητος είναι ο μηχανισμός συλλογής των κονδυλίων. Εξακολουθώ να θεάρα εαυτόν ε, ε, ως ένα πολιτικό ο οποίος βασίζεται σε στοιχεία και Ο Επίτροπος λέει πως όλα τα ποσά μέχρι 5.000 ευρώ δεν θα περικοπούν κάτι το οποίο ακούγεται λογικό, αλλά μετά βεβαίως έχει το εξής αποτέλεσμα. Στις χώρες, στα κράτη-μέλη θα υπάρξει μια τεράστια ανισορροπία. Είναι ακατανόητο να επιτρέψουμε κάποιες χώρες λόγω της δομής των εκμεταλλεύσεων δεν θα α, συνεισφέρουν τίποτα. Παραδείγματος χάρη η Γαλλία πρέπει να πληρώσει τόσα όσα και η Πολωνία για τον Αραβόσιτο. Πώς το εξηγούμε αυτό ή επίσης για ποιο λόγο να κάνουν οικονομίες οι αγρότες ε, όταν αυτό δεν ωφελεί σε τίποτα ή τουλάχιστον δεν ωφελεί αναλογικά Οπότε η έκθεση αυτή ε, είναι και κάπως αντιφατική. Το δικαιότερο σύστημα είναι, αν χρειάζεται λεφτά ο προπολογισμό των ε, Βρυξελών, να κόψουμε από την ε, γραμμή Α για την δημοσιονομική πειθαρχία. Οι προτάσεις ε, που ακούστηκαν δεν ε, θεωρώ πως είναι μια συνεκτική πολιτική. Και θεωρώ πως θα πρέπει να υπάρχει, όπως είπα, μια ομοιόμορφη εφαρμογή. Και από αυτό προκύπτει πως ε, θα, υπάρχει, θα υπάρχουν λιγότερες περικοπές σε όλες τις χώρες και αποτελεσματικότερη χρήση του προϋπολογισμού. Αν σκεφτούμε πως στη νέα περίοδο προβλέπονται περισσότερες δαπάνες, τότε ο μηχανισμός αυτός δημοσιονομικής ταρχίας θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία. Γι' αυτό θεωρώ πως όλες οι χώρες Ευρώπης θα πρέπει να συμμετάσχουν επίσης όρες. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ντεκάστρο για ένα λεπτό. Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, να το πω με σαφήνεια και στεναρά. Δεν μπορεί να δοθεί την περικοπή των άμεσων πληρωμών ε, το Κοινοβούλιο, όπως τις έχει περιγράψει τα συμπεράσματα από το Συμβούλιο στις 7 τον 7 και 8 Φεβρουαρίου. Θα πρέπει να δοθούν τα δικαιώματα που αρμόζουν στο Κοινοβούλιο, όπω προβλέπουν και οι συνθήκε. Ω θεσμικό όργανο, με την μέγιστη δημοκρατική διαφάνεια, θα πρέπει να προβλέψουμε ένα σύστημα συνεπέ για του Ευρωπαίου δικαιοργού. Εν αναμονή συμφωνία, λοιπόν, η παρακοπή των άμεσων πληρωμών θα πρέπει να βασιστεί στο ανώτατο όριο για το 2014, όπω το έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή τη για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό είναι συμβατό και με τη δημοκρατική εντολή που έχει εγκρίνει η Ολομέλεια για τον κανονισμό των άμεσων πληρωμών. Επιπλέον, η Επιτροπή Γεωργίας, όπου προεδρεύω, έχω την τιμή να προεδρεύω, δεν θεωρεί ότι όλοι οι γεωργοί θα πρέπει να τιμωρηθούν με το ίδιο ποσοστό περικοπή, ανάλογα, άσχετα μάλλον με τι διαστάσει των εκμεταλλεύσεων του και το τι βοήθεια λαμβάνουν. Δεν μα φαίνεται ούτε δίκαιο ούτε λογικό, γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να του στηρίξουμε. Αυτοί που λαμβάνουν έω 5.000 ε, ευρώ βοήθεια θα πρέπει να στηριχθούν. Ευχαριστούμε. Για δύο λεπτά κυρία Ράιμερς. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχει ολοκληρωθεί το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ακόμα δεν έχουμε ε, κερδίσει τον σεβασμό του Ευρωπαίου πολίτη που υποτίθεται ότι εκπροσωπούμε. Τώρα, με βάση εκτιμήσεις πρέπει να αποφασίσουμε και τα δεδομένα αυτά απαιτούν, λέει, περικοπή του προϋπολογισμού της γεωργίας. Εδώ πέρα πρέπει να υπάρχει λοιπόν ισονομία. Όλοι οι γεωργοί έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Οπότε θα πρέπει εδώ πέρα να θα πρέπει να υπάρξει μια οριζόντια περικοπή για ε, να έχουν όλοι νομίζω την ίδια υπευθυνότητα στην ε, χρήση των χρημάτων. Δεν είναι δυνατόν στην Ευρώπη να γίνεται η μόδα ε, να σκεφτόμαστε με άσπρο και μαύρο και να λέμε αν οι δομές είναι μεγάλες ή μικρές. Αυτό είναι λάθος, επικίνδυνο και επικίνδυνο και για την ευρωπαϊκή σκέψη, γιατί πρέπει από κοινού να ε, καταλήξουμε σε έναν στόχο. Και ε, από κοινού να σηκώνουμε και τα βάρη. Οπότε πρέπει να είναι οριζόντια η περικοπή, να μην εξαιρεθούν τα ποσά κάτω από 5.000 ευρώ και οι μικρές εκμεταλλεύσεις. Πρέπει να μάθουν πως ε, σε βάθος χρόνου θα υπάρχουν λιγότερα λεφτά. Και άμα το ξέρει κανείς θα κάνει και τα κουμάντα του. Δεν έχει νόημα να ε, νομίζουν οι μικρές εκμεταλλεύσεις πως θα παραμείνουν τα πράγματα τα ίδια. Όχι. Θα φέρουμε τους αγρότες σε σύγκρουση και προωθεί, όπως είπα, αυτή τη λογική του άσπρου μαύρου. Και δεν είναι σωστό αυτό για μια έτσι πανευρωπαϊκή σκέψη. Σας ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κάπουλα Σάντος ε, που ανέλαβε αυτή την έκθεση εν το μέσο τεταμένων διαπραγματεύσεων. Πραγματικά δηλαδή είναι μαζόχας. Φαντάζομαι πως είχε αρκετή δουλειά χωρίς και αυτή την έκθεση. και χωρίς να ασχολείται με τα γεωργικά. Οι συνολικές δαπάνες ε, της κοινή γεωργικής πολιτικής έχουν φτάσει σε τέτοιο μέγεθος που πρέπει να υπάρξει κάποια πειθαρχία για να παραμείνουμε εντός των πλαισίων ε, των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, από ό,τι φαίνεται όμως πως η Επιτροπή, η Επιτροπή Γεωργίας υπολογίζει ένα ποσοστό προσαρμογής και κατόφλι που θα έχει δυσανάλογα αποτελέσματα για πολλούς αγρότες. Το κατόφλι των 5.000 ευρώ που προτείνεται σημαίνει πως 80% των αγροτών εξαιρούνται. Mm. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, αλλά εγώ δεν μπορώ να δικαιολογήσω σε οποιονδήποτε ψηφοφόρο μου αγρότη το ότι 20% θα πληρώσουν, 20% ε, από αυτούς μόνο θα πληρώσουν το έλλειμμα που αντιστοιχεί σε όλα τα κρατημέλη και όλους τους αγρότες. Πρέπει να υποστηρίξουμε ένα μέτρο το οποίο οπωσδήποτε Ε, δεν θα οδηγήσει σε τέτοιες ανισότητες μεταξύ κρατών μελών και αγροτών και οπωσδήποτε καταστρέφει οποιαδήποτε ελπίδα ίσων όρων ανταγωνισμού. Ο κανονισμός αυτός είχε στόχο να διασφαλιστεί πως το βάρος θα το μοιραστούν εξίσου και δίκαια όλοι οι αγρότες στην Ένωση. Αυτό πρέπει να κάνουμε κύριε Πρόεδρε και αυτό πρέπει να κάνετε εσείς, κύριε Επίτροπε. Η δε πρότασή σας είναι άδικη, ανεπαρκής και απαράδεκτη. Ευχαριστώ. Κύριο Σομαρζή για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, με εκπλήσει κάπως η εφαρμογή που ζητάτε του κανονισμού αυτού στις απομακρυσμένες περιοχές και στις νήσους του Αιγαίου αφού τους εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες. Αν κατάλαβα καλά, του ζητάτε τώρα να συμμετάσχουν στην ε, χρηματοδότηση ενός αποθέματος κρίσεως που με το οποίο δεν θα μπορούν να υποφεληθούν. Δεν μπορούμε επίσης να γνωρίσουμε ότι η μείωση που προβλέπει ο κανονισμός θα μεταφραστεί σε μείωση των ποσών που θα διατεθούν και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές για το 2013, αντίθετα από τις δεσμεύσεις που είχαν αναλυφθεί. Ξέρω κύριε Επίτροπε ότι επιμένετε οι ιδιαιτερότητες αυτών των περιοχών να ληφθούν υπόψη και γι' αυτό κατατίθεται η τροπολογία 2 με άλλους 40 συναδέλφους δηλαδή ώστε ο κανονισμός αυτός να μην εφαρμοστεί στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές και στις νήσους του Αιγαίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό κύριο Στογιάννο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Положението на Европа на Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, το πρόβλημα εδώ πέρα είναι το εξής. Τα παλιά κράτη-μέλη είναι σε προνομιακή θέση, τα νέα και μικρότερα παραμένουν αβοήθητα. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί να μην παίρνει ο Πολωνός αγρότης όσα παίρνει και ο Γάλλος. Και μας λέτε δεν μπορώ να το εξηγήσω στους Γάλλους αγρότες. Στους Πολωνούς αγρότες δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε, στους Βούλγαρους αγρότες. Δηλαδή πόσο καιρό ακόμα θα ανεχόμαστε αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η ενωμένη στην πολυμορφία. Σας στάνει τόση πολυμορφία ή θέλετε κι άλλοι. Εδώ πέρα πλέον έχουμε φτάσει σε καταστάσεις ε, φάρμας των ζώων. Κάποιοι είναι πιο ίσοι από του άλλου. Ντόφμαν. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι λυπηρό το ότι συζητάμε καν αυτό το θέμα. Γιατί τα τελευταία χρόνια δεν τηρήσαμε τα επεσχημένα και δεν υπάρχει άρα ασφάλεια δικαίου για την 7 προγραμματική περίοδο. Αλλά κάνατε μια πρόταση κύριε Επίτροπε για πώς θα γίνουν οι περικοπές. Και νομίζω πως είναι ένα μικρό σημάδι προς την κατεύθυνση της στήριξης των μικρών επιχειρήσεων. Δεν μιλάμε για μεγάλα νούμερα. Κατά μέσο όρο μιλάμε για 10-15 ευρώ ένα εκτάριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει νόημα νομίζω, είναι σωστό. Εάν είναι να επιζήσουν οι μικρές εκμεταλλεύσεις πρέπει και εμείς να δώσουμε ε, τα μηνύματά μας. Αλλά πάει προς σωστή κατεύθυνση. Βεβαίως είναι ζήτημα κατανομής μεταξύ κρατών μελών. Και εδώ πέρα συμφωνώ με τον συνάδελφο πως έπρεπε να το έχουμε λύσει διαφορετικά να καθοριστεί κάτι στα κράτη-μέλη ως περικοπή και μετά το κράτος μέλος να αποφασίσει τι θα κάνει. Δεν συνέβη αυτό, τέλος πάντων. Η πρόταση αυτή για τις ε, μικρές ε, εκμεταλλεύσεις ε, είναι σωστή. Γι' αυτό και θα υποστηρίξω την πρότασή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκαρσία Πέρες για ένα λεπτό. Πρόεδρε, Επίτροπε, ο Ισπανός Υπουργό Γεωργίας, Κανιέτε, ανακοίνωσε θριαμβευτικά ότι η συμφωνία αυτή ήταν πολύ θετική, διότι δεν θα επιφέρει μειώσεις στην γεωργική πολιτική της Ισπανίας. Οι συνέπειες όμως δεν θα είναι ακριβώ αυτέ. Εξαρτάται από το σχέδιο κανονισμού τη δημοσιονομική πειθαρχία. Όπω το υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για, για το πολιτή δημοσιονομικό πλαίσιο. Προβλέπει μάλιστα άμεση περικοπέ στι άμεσε πληρωμέ για του γεωργού τη δική μα περιφέρεια. Ε, η σοσιαλιστική λοιπόν αντιπροσωπεία του σώματο δεν είναι καθόλου υπέρ αυτή τη ε, Είμαστε κατά τη περικόπη που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει τη συμφωνία που ω τώρα έχει γίνει. Το Συμβούλιο θέλει να επιφέρει περικοπές σε στις τι ε, πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωση. Δεν μπορεί λοιπόν το Κοινοβούλιο να συμφωνήσει ακόμα σε αυτό. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό κυρία Όγιουλαντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κανονισμό για τη δημοσιονομική επιθαρχία σκοπό έχει να διασφαλίσει ότι οι επικαλύψει και επαναλήψει τη άμεση πληρωμέ θα γίνονται σεβαστέ Δυστυχώ όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πάει ακόμα μακρύτερα και ζητά πλέον μέσο αγοράς οι οποίες να διασφαλίζονται και να χρηματοδοτούνται από τον προπολογισμό της ΚΑΠ. Η σοβαρή περικοπή για τους ε, άμεσες ενισχύσεις των γεωργών που λαμβάνουν 5.000 που λαμβάνουν άνω των 5.000 ευρώ θα σημαίνει μια μείωση δισεκατομμυρίων ευρώ, τουλάχιστον 5 Ε, κάτι που είναι το διπλάσιο ποσό από αυτό που θέλει να καλύψει αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταλαβαίνω ότι θέλουν να εξοικονομήσουν στο δυνατόν περισσότερα από κάθε δημοσιονομική γραμμή, αλλά αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πάει πάρα πολύ μακριά. Θέλω λοιπόν να καλέσω του συναδέλφου να στηρίξουν τον ε, εισηγητή και την αρχική πρόταση τη Κομισιόν. Την αρχική να περικοπούν κατά 0,7% οι άμεσε πληρωμέ και να συμπεριλαμβάνονται μόνο οι γεωργοί που λαμβάνουν άνω των ε, 5.000 ευρώ. Δεν συμφωνώ με τι τιμέ τη αγορά και το σχετικό αποθεματικό. Όμω αυτό θα πρέπει να συντίθεται από διαφορετικά ταμεία και διαφορετικού πόρου. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριο Σάιμον. Ευχαριστώ κύριε και κύριοι. Θα ήθελα να δηλώσω ρητά ότι δεν υποστηρίζω την πρόταση της Κομισιόν για τις επιλεκτικές περιοκοπέ στις άμεσες πληρωμές για τους γεωργούς το 2013. Το θέμα είναι εάν αυτή η πειθαρχία, αυτά τα πειθαρχικά μέτρα είναι απαραίτητα σε αυτή τη φάση. Λόγω του ότι δεν υπάρχει πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 14 με 20, δεν υπάρχει και λόγος να γίνουν αυτές οι περικοπές. 5% στις άμεσες πληρωμές. Εγώ υποστηρίζω την πρόταση του εισηγητή ότι το 1% θα αρκούσε και αυτό θα υποστηρίξω αύριο στην ψηφοφορία. Το χειρότερο είναι η επιλεκτικότητα αυτών των περικοπών. Η προσέγγιση της Κομισιόν μιλάει για 5.000 ευρώ. Δηλαδή οι μικροί γεωργοί δεν θα χρειαστεί να σφίξουν το ζωνάρι τους, μόνο οι, μικρο, οι μεσαίοι και οι μεγάλοι. Αυτό είναι κάτι που δεν με βρίσκει σύμφωνο. Πρέπει να υπάρξει περικοπή για όλους και αν δεν γίνει κάτι τέτοιο τότε θα, υπά, θα δοθεί άδικη θα υπάρξει άνηση μεταχείριση για τους Τσέχους γεωργούς αυτό είναι απαράδεκτο δεν χρειάζεται να σκεφτούμε τη φάρμα των ζώων ξανά για δύο λεπτά μάτο αντρόβερ Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Η εξαίρεση ορισμένων από την πειθαρχία που προβλέπει η πρόταση είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνουν οι γεωργοί. Η Κομισιόν προτείνει μείωση 14 και μισών εκατομμυρίων πράγμα το οποίο θα δυσχεράνει τη ζωή ορισμένων περιφερειών και όλων όσων εξαρτώνται από την ΚΑΠ. Ήδη είχε εγκριθεί μια τροποποίηση και το Κοινοβούλιο ήθελε αύξηση των ταμείων για τις απομακρυσμένες περιοχές που δεν έχουν αρκετή στήριξη. Η Γαλλία, η Ισπανία εδώ και χρόνια χορηγούν επιχορηγήσεις και βοήθειες και στηρίξεις για να συμπληρώσουν ό,τι τους δίνει η ΚΑΠ. Οι ζώνες αυτές οι απομακρυσμένες πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση με έχουν ανεργία πάνω από 50% και όπως είχε γίνει και σε άλλες περιπτώσεις με βάση το 349 της συνθήκης πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιδείξει αλληλεγγύη με αυτούς τους γεωργούς των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιοχών. και να του τύχουν ιδιαίτερες μεταχείρισης. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, ο κύριος Ανδριού. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Λουίς Μανουέλ Καπόλας Σάντους για το έργο του και την έκθεση του προφανώς τη στηρίζω. Στην πραγματικότητα αυτά που αναφέρεται επίτροπε είναι μία πλευρά της πραγματικότητας. Αλλά από την άλλη το Κοινοβούλιο είναι μέλος διαδικασίας της συναπόφασης και είναι σύνομο θέτης βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας. Η πρόταση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενώ δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι απαράδεκτη διότι μας ζητάτε να αποδεχτούμε ένα ποσοστό αναπροσαρμογής των ε, άμεσων πληρωμών της ΚΑΠ για το 2014 βάσει το 2013 με μείωση του 0,5% κάτι μου φαίνεται απαράδεκτο έτσι όπως έχει. Ε, η ιδιαιτερότητα των εξόχως απομακρυσμένων περιοχών και των εκμεταλλεύσεών τους όπως τις καλύπτει και η συνθήκη. Είναι στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ε, για αυτό το σκοπό και σήμερα και αύριο θεωρώ ότι θα πρέπει να μην γίνουν ε, μειώσεις κατά κανένα τρόπο στις εκμεταλλεύσεις αυτών των ευάλωτων περιοχών και περιφερειών. Πρόεδρος, ευχαριστούμε και τώρα να ξεκινήσουμε τη διαδικασία Catch the Eye. Δύο μιλητές. Πρώτα απ' όλα κύριος Δανέλης. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καλώ και εγώ τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν τις τροπολογίες που υποστηρίζουν την εξαίρεση των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τη γραμμική μείωση που ενδεχομένως χρειαστεί να επιβληθεί μετά την οριστικοποίηση του προϋπολογισμού για την περίοδο 2014-2020. Ας μην ξεχνάμε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι δεν είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις αυτές που επιβαρύνουν με το μερίδιο του λέοντος τον προϋπολογισμό για τις άμεσες ενισχύσεις. Αντίθετα, στις μικρές εκμεταλλεύσεις οφείλεται η προσφορά πληθώρας κοινωνικών αγαθών, τα οποία δεν ανταμείβονται από τις αγορές ένα τέτοιο αγαθό είναι και η αντίσταση στην απερίμωση απομακρυσμένων περιοχών οι οποίες ούτως ή άλλως βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. γι' αυτό το λόγο και ζητάμε επιπροσθέτως την εξαίρεση από τη μείωση και των μικρών νησιών του αιγαίου καθώς και των εξόχως απόκεντρων περιοχών. σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά πρώτον, να πω στον Επίτροπο ότι ελπίζω και εκείνος και η Ιρλανδική Προεδρία να βρουν επιτέλους κάποια λύση. Να βρουν μια λύση σε ό,τι αφορά την κοινή αγροτική πολιτική πριν το τέλος της Ιρλανδικής Προεδρίας, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αν γίνεται. Αν τα καταφέρουμε, θα έχουμε επιτύχει κάποια πρόοδο και μάλιστα ουσιαστική. Εάν μπορέσουμε μάλιστα να μεταφράσουμε αυτή την πρόοδο στην νομοθεσία, θα τα έχουμε πάει και καλά. Σε ό,τι αφορά την έκθεση που συζητούμε απόψε το βράδυ, δεν είναι απλό. Ούτε ευχάριστο για όλους τους μπλεκόμενους και τους ενδιαφερομένους αυτό που συμβαίνει. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι αναθεώρηση. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και πρέπει να είμαστε και πραγματιστέ. Και αν θέλουμε να είμαστε πραγματιστέ, αλλαγέ χρειάζονται. Αλλά θα πρέπει να γίνει και εξαίρεση για τι μικρέ εκμεταλλεύσει. Όχι μόνο γιατί αυτέ εξαρτώνται από τι συγκεκριμένε άμεσε πληρωμέ, αλλά γιατί πραγματικά είναι θέμα επιβίωση για αυτέ τις συγκεκριμένη εξαίρεση. Πρόεδρο, ευχαριστώ να δώσω το λόγο στον Επίτροπο Τσιόλο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τώρα θα μπορέσω να επαναλάβω κάποια στοιχεία και να αποσαφηνίσω. Η πρόταση αυτή, κύριε Αντριέ, δεν έχει να κάνει με έλλειψη σεβασμού κατά του Κοινοβουλίου. Είναι ένα μέτρο προφύλαξης. Εάν το Κοινοβούλιο φτάσει στο τέλος των διαπραγματεύσεων για τις δημοσιονομικές προοπτικές με το Συμβούλιο και καταφέρει να αυξήσει τον προπολογισμό της ΚΑΠ και να φτάσει στο επίπεδο της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκή Επιτροπής δεν θα υπάρξει λόγο να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό. Προ στιγμήν όμω, οι αριθμοί που έχουμε μπροστά μα και έπειτα από ήδη υπάρχουσα απόφαση του Συμβουλίου είναι οι αριθμοί ακριβώ αυτοί. Αντί λοιπόν τώρα να έχουμε μια μικρή μείωση και να υποχρεωθούμε μετά από λίγους μήνες να επιφέρουμε μεγαλύτερε δραστικότερε μείωσει. καλύτερα είναι να το πάρουμε τώρα αυτό το μέτρο, το προφυλακτικό, διότι πρόκειται το ή για νομοθετική πρόταση. Εσεί αποφασίζετε τι θα κάνετε έτσι κι μαζί με το Συμβούλιο, το διευκρίνησα και προηγουμένω. Το ε, διευκρίνησα, μπορούμε με το διορθωτικό προπολογισμό να επανέλθουμε. Να επανέλθουμε στη μείωση που είχαμε προτείνει αρχικά και έτσι να μειωθεί λιγότερο το ποσοστό των άμεσων πληρωμών. Δεύτερο, στοιχείο για να απαντήσω. Λέτε ότι παίρνουμε τα χρήματα των γεωργών. Η δημοσιονομική πειθαρχία εφαρμόζεται μόνο για τις περιπτώσεις το Ταμείο της Κρίσης που παραμένει εντός της ΚΑΠ για τους γεωργούς. Οι γεωργοί θα είναι οι δικαιούχοι. Αλλά δεν, μπορούμε να, δεν να λέμε ότι παίρνουμε τα χρήματα των γεωργών από την ΚΑΠ και τα πάμε αλλού, κάπου άσχετα. Κυρία Γκερσέπερες, θα θυμάστε, πριν από δύο χρόνια νομίζω, είχαμε κρίση στον τομέα των οπορκυπευτικών. Και επειδή υπήρχε το ταμείο αυτό για την αντιμετώπιση τη κρίση, μπορέσαμε να βοηθήσουμε την Ισπανία και έτσι καλύψαμε του παραγωγού οπορκυπευτικών. Έτσι καλύψαμε ένα μέρο των απολειών του λόγω τη κρίση. Αυτά είναι τα χρήματα που μαζεύουμε. Δεν πετιούνται. Δημιουργούμε ένα ταμείο για την αντιμετώπιση τη κρίση και αν δεν χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια στο 2014 ε, για σκοπού αντιμετώπιση κρίση, εφόσον δεν υπάρξει κρίση, δεν θα χαθούν. Στα χέρια των Γεωργών θα πάνε έτσι κι αλλιώ. Αποθεματικό λέγεται. Γι' αυτό το σχηματίζουμε και πάντοτε δικαιούχοι θα είναι Γεωργοί. Ε, τώρα, για τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Κύριε Νίκολσον, έχετε δίκιο. Μιλάμε για το 80% των γεωργών που θα εξαιρεθούν. Αλλά θα θυμάστε ότι το 80% των γεωργών λαμβάνουν μόνο 20% των άμεσων πληρωμών. Οπότε, εξαιρούμε τους γεωργούς που συνολικά παίρνουν 20% των άμεσων πληρωμών. Δεν μπορώ λοιπόν να σας αφήσω και με την εντύπωση ότι μόνο ένα μικρούλι μέρος των γεωργών είναι υπέρ αυτού του μέτρου. Είναι μικρότερο μέρος με των γεωργών, αλλά λαμβάνουν μεγάλο μέρος των πληρωμών. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα μέτρο δίκαιο. Όχι από διοικητικής άποψης μόνο είναι απλούστερο, διότι με το όριο των 5.000 αυτό μειώνουμε κατά 80% το διοικητικό άχθος, αλλά επικεντρωνόμαστε και σε αυτούς που παίρνουν τις μεγαλύτερες πληρωμές. Για τον κύριο Ποζέ να για τα ποζέι μάλλον, για τις περιοχές ποζέι, να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σέβεται αυτά που έχει πει ο νομοθέτης. Ο ισχυρός κανονισμός προβλέπει ότι η διαφοροποίηση δεν εφαρμόζεται στις περιφέρειες ποζέι, όμως η δημοσιονομική πειθαρχία ισχύει για αυτές. Τι θα πει αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε την επιλογή. Δεν είχε επιλογή γιατί έπρεπε να σεβαστεί του κανόνε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει προτάσει νομοθετικέ, λαμβάνοντα υπόψη κάποιου κανόνε οι ίδιοι κανόνες που λένε ότι για να, για εφαρμοστεί η συναπόφαση θα πρέπει το Συμβούλιο και η Επιτροπή να λάβουν απόφαση στις 30 Ιουνίου. Η απόφαση αυτή, εάν δεν ληφθεί, τότε θα ισχύει ο... Υπάρχουν δημοσιονομικός κανονισμός που προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αργότερα θα υποβάλει την πρότασή τη. Αυτέ ήταν οι εξηγήσει που ήθελα να δώσω. Νομίζω ότι τα πράγματα τώρα είναι σαφέστερα. Και ελπίζω να είχατε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να λάβετε την αποφασή σα. Εν πλήρη γνώση τη κατάσταση. Πρόεδρο, ευχαριστούμε, Επιτροπέ, για αυτή την απάντηση. Τελευταίο ομιλητή, ο κ. Κάπολα Σάντου. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ο Επίτροπος έχει δώσει πάντοτε δείγματα εξαιρετικής συνεργασίας με το Κοινοβούλιο. Και πραγματικά καταγράφουμε με εκτίμηση την προθυμία του να υπάρξει διάλογος μαζί μας. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για την Επιτροπή συνολικά σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι υπάρχει πραγματισμός ή ρεαλισμός πολιτικού χαρακτήρα που να διακυβεύει την ε, ισορροπία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Για αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι η στάση ως προς το θέμα αυτό θα έπρεπε να μεταβληθεί. Το επαναλαμβάνω. Και θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις ε, εισηγήσεις τους, διότι θα ενισχυθούν έτσι περαιτέρω οι αρχικές θέσεις του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ για την έγκριση του περιεχομένου τη έκθεση. Δείχνουν έτσι τη συνεπή του στάση οι βουλευτέ, δείχνουν ότι σέβονται την εντολή που έχουν αναλάβει από του πολίτε και επανεπιβεβαιώνουν το ότι υπερασπίζονται πάνω από όλα τα δικαιώματα των γεωργών. Των γεωργών και αυτό για το μεγαλύτερο μέρο των συναδέλφων. Και μάλιστα υπερασπίζονται του μικρότερου γεωργού. Σα ευχαριστώ όλου. Κλείνει η συζήτηση. Ψηφοφορία αύριο στι 11.30. Κυρίε και κύριοι, επόμενη συνεδρίαση αύριο. 12 Ιουνίου 2013 στις